Not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 Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Ε, Μόλον ότι απουσιάζουν πολλοί συνάδελφοι, πάντω γιατί ο χρόνο τρέχει. Θα σα ενημερώσω σχετικά με τα αποτελέσματα τη συνεδριάσεω των ε, συντονιστών σήμερα το πρωί. Ξεκινήσαμε με το διορισμό των εισηγητών και των ε, εισηγητών γνωμοδοτήσεων. Λοιπόν, προτείνεται να συνταχθούν το παρακάτω. Μια έκθεση για το DCI και θα αναλαμβάνει αυτή την έκθεση το ELK Έκθεση πρωτοβουλίας, όπως είσαμε για τις παρακάτω εκθέσεις, επί ανακοινώσει τη Κομισιόν για την συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης, δημιουργίας ενός πολιτικού πλαισίου για το θέμα της αιτήσεις ε, ανάπτυξη και τίτλος της, της ε, έκθεσης θα είναι η συνοχή των ε, πολιτικών για την ανάπτυξη και οι πράσινοι θα την αναλάβουν. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συνένεσης επί, της, επί ζητημάτων ανάπτυξης είναι το ΕΛΚ που θα την αναλάβει. Αποφασίσαμε να μην συντάξουμε εκθέσεις για τα παρακάτω θέματα επί τη ανακοινώση τη Κομισιόν για την ε, σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Λατινική Αμερική, ζητάμε να αποκτήσουμε το καθεστώς ε, συνεργαζόμενης επιτροπής εάν λάβει κάποια άλλη κοινοβουλική επιτροπή μια έκθεση το θέμα της έδρας της ε, Νάπολης ως έδρα της συνέλευσης. Ε, θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι κάτι το που αντιβαίνει στις ρυθμίσεις ε, του Κοτονού. Έχουμε ήδη αποφασίσει να συντάξουμε γνωμοδοτήσει. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Λίμπε θα αποφασίσει να συντάξει έκθεση επί των κανονισμών του κανονισμού για ορισμένα περιοριστικά μέτρα προς την Σομαλία και την Ζιμπάμπουε για τη Σομαλία είναι ε, για τη Σομαλία θα το αναλάβει το ΕΛΤΟ σε ό,τι αφορά τις ομάδες εργασίας και τους ε, ειδικού ηγητές ομάδα εργασίας για τις ε, νομοθετικά μέσα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΔΕΒΕ οι συντονιστές έχουν βεβαίωσει την ε, σύσταση πέντε ομάδων εργασίας και σας ότι αυτές οι ομάδες ε, προεδρεύονται από τον Νόρμπερ Νόιση, ομάδα Β από τον Νίρ Σουντέβα, ομάδα Γ από τον Δαβίδ Μαρία Σασόλη, Ντε Γκέρενς και Ε Μισελ Στριφλέρ. Οι ομάδε που δεν έχουν ακόμα ορίσει τους εκπροσώπου της ομάδα. παρακαλώ να το πράξουν άμεσα και τα τακτικά μέλη προηγούνται για την ε, ανάθεση εκθέσεων. Επίσης ε, διορίσαμε μέλη τα οποία συμμετέχουν στην ομάδα Ασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένα Έθνη, τέσσερα μέλη. Καθένα από τα μέλη των ομάδων ΠΕΠΕ, και ΑΛΔΕ θα ορίσουν στο μέλλον τα, τους εκπροσώπους τους τώρα για μια έκθεση σχετικά με τη σχέση με την, Ευρωπαϊκή με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν προωθήθηκε. Θα κάνουμε κάποιες ε, ακροάσεις το 2010 και προτείνεται να ε, να οργανώσουμε τις παρακάτω ακροάσεις. Ακρόαση για την κατάσταση στην Παλαιστίνη, κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Αλίας για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της Αλίας, ακρόαση για προβλήματα της ε, έγκυας ιδιοκτησίας στις αναπτυσσόμενες χώρες που θα εξετάσουν επίσης και τα θέματα της κατάσχεσης γεών και το θέμα της ε, απειλής ε, για την επιστημική ασφάλεια και έδωσε επίσης ε, και μια ακρόαση για τα παιδιά. Μπορούσαμε επίσης να σας προτείνουμε κάποιες αντιπροσωπείες της Επιτροπής μας το 2010 Έχουμε φέσει για τις εξή περιοχές, Παλαιστίνη, Νότιο Σουδάν, Βόρειο, Βόρεια Κένια, για να εξετάσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση και την Βραζιλία, μεταξύ άλλων τα προβλήματα της ε, καταπάτησης των γεών. με αυτές τις επιτροπές ad hoc για την τρίτη διάσκεψη Ευρώπης, Αφρικής, Λιβύης για τους και για, το στόχου της Επίσης ε, έχουμε κάποια απομεινάρια από χρήματα θα λέγαμε, υπολείμματα, γι' αυτό να εξετάσουμε, να κάνουμε δύο μελέτες για τις διακρίσεις στην βοήθεια για ανάπτυξη και δεύτερον η πολιτική δάστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εταιρική σχέση, μάλλον σύμπραξη δημόσιο ιδιωτικού τομέα και επίσης έχουμε ορίσει άτομα που θα εδρεύουν στο εκτελεστικό συμβούλιο και τα τακτικά μέλη είναι Σνίμπερ για Στραμ και ο Μαρτίνες και αναπληρωματικά μέλη Τσίμερ και Γκέρτς. αποφασίσαμε να προτείνουμε την κατάρτιση προφορική ερώτηση για την ε, σεξουαλική βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Και αυτό αφορά στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αιτήματα που έχουμε λάβει, οι συντονιστές ε, προτείνουν να γνώσουμε τα παρακάτω, τις παρακάτω διοργανώσεις ε, για τη σημασία των φόρων και των δασμών στις αναπτυσσόμενες χώρες που θα διοργανωθεί το 2009. Και συνάντησα τον, Υπουργό, τον Επίτροπο Ντεγκούχτ και πιστεύουμε να διεξαχθεί αυτό το, αυτή η εκδήλωση αρχές Δεκεμβρίου. Το η δημιουργία ενός ε, ενός ε, χώρου που θα εξετάζει διάφορα ανθρωπιστικά ζητήματα. Θα οργανώσουμε μια συζήτηση με τους ε, εμπειρογνώμονες σε θέματα παροχής βοήθεια. Ε, όλα τα υπόλοιπα αιτήματα πέρασαν, θα περάσουν μέσω γραπτή διαδικασία. Συμφωνείτε με τις συστάσεις των συντονιστών. Ωραία. Και τώρα να σας κάνω μια ανακοίνωση. Αύριο θα ψηφίσουμε της ε, σύστασης ειδική Επιτροπής ε, για την ε, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και υπάρχει συγκεκριμένη εντολή για την Επιτροπή αυτή. Μετά από την ανάγνωση του κειμένου, μάλλον εντολής, θα ήθελα να πω ότι μας εκπλήσει το γεγονός ότι η εντολή που ανατίθεται σε αυτήν την ειδική επιτροπή δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την κρίση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω την άδεια να προτείνω δύο προφορικές τροπολογίες αύριο κατά τη διάρκεια ψήφισης αυτού του κειμένου έτσι ώστε και τα συμφέροντα των αμφισωμένων χωρών να συμπεριληφθούν. Συμφωνείτε? Σας ευχαριστώ. Σημείο 16 της Διατάξεως που είναι η έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος για το 2010. Το έχετε όλοι. θα να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Εγκρίθηκε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Είναι εδώ η προσκεκλημένη μας. Ωραία. Θα εξετάσουμε λοιπόν την κατάσταση τώρα στην Μαυριτανία. Μετά από το πραξικόπημα ξεκίνησαμε διαβούλευση στο πλαίσιο του άρθρου 96 Συμφωνίας Κοτονού και η Επιτροπή είχε διακόψει την ε, Συμφωνία Συνεργασίας στο το πλαίσιο, υπήρξαν εκλογές το 2009, τις οποίες ε, κέρδισε ο επικεφαλής ε, του πραξικοπήματος. Υπάρχουν ισχυρισμοί περί νοθείας ε, και καταγγελίες. Ε, γι' αυτό θελήσαμε να ακούσουμε λοιπόν την Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να μας ενημερώσουν περί της καταστάσεως στην Μαυριτανία. Να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρούνο Κάτα, εκ μέρους Επιτροπής. Merci Madame la Présidente. Comme vous venez de le rappeler, la Mauritanie... Όπως μόλις το θυμήσατε, η Μαυριτανία βρίσκεται σε φάση διαβούλευση στα πλαίσια του άρθρου 96 της συνθήκης του Κοτονού και αυτό λόγω του πραξικοπήματος το 2008 και οι διαδικασίε του άρθρου 96 άρχισαν, ε, ενισχύουν τον Απρίλιο του 2009 με την επιβολή κυρώσεων. Δηλαδή σταμάτησε η χρηματοδότηση μέσα στα πλαίσια του 10ου ΦΕΔ και μερικών υπολοιμάτων του παρελθόντος για ένα σύνολο των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από διαπραγμάτευση με μεσολαβητή τις αρχές της Ενεγάλης και τον πρόεδρο Ατμάχ, επήλθε συμφωνία η οποία οδήγησε στις εκλογές που μόλις αναφέρατε. Η συμφωνία οδήγησε στην αποδέσμευση ενός πρώτου μερικού ποσού της συνεργασίας και μετά τις εκλογές αποδεσμεύτηκε ένα άλλο ποσό, δηλαδή 230 εκατομμύρια δόθηκαν και 136 εκατομμύρια είναι ακόμα μπλοκαρισμένα περιμένοντας τις εξελίξεις. Οι εκλογές αποτελούν καρπό της συμφωνίας. Δεν έχει γίνει επαλήθευση για το πόσες απάτες έχουν γίνει και νοφίες. Πάντως, έχουμε τώρα μία μεικτή αποστολή Κομισιόν Συμβουλίου που στα πλαίσια του άρθρου 96 πήγε να διαπιστώσει πώς έχει κατάσταση στη Μαυριτανία και κατά πόσο οι συμφωνίες του Ιουνίου 2009 γίνονται σεβαστές. Ακόμη η αποστολή βρίσκεται επί τόπου και θα αναφέρει το συντομότερο στο Συμβούλιο. Και ανάλογα με το τι συμπεράσματα θα βγάλει αυτή η Επιτροπή, η Ερευνητική Επιτροπή, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε στη συνέχεια για τις κυρώσεις. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψει η αποστολή από την Μαυριτανία και να μας πει τα καθέκαστα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Γιώχαν Νίλσε από το Συμβούλιο για να μας πληροφορήσει σχετικά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι το βασικό σημείο είναι οι αποστολή σύμφωνα με το άρθρο 96, οι οποίε βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ όσο μιλάμε. Σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να προδικάσουμε τα αποτελέσματα από αυτή της αποστολής. Όπως είπε και ο Μπρούνο Γκάτα, η ε, Κομισιόν ε, εξετάζει τις εξελίξεις και περιμένει να γίνουν συζητήσεις με τους βασικούς ε, πολιτικούς πρωταγωνιστές. Λοιπόν, ε, παραλαμβάνω ότι η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το 96, και ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα στις Βρυξέλλες με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Euh, Θέλει κανείς ε, να ρωτήσει κάτι. Όχι. Πάμε στο επόμενο σημείο. Είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό. πρόκειται για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συζήτηση επαναργάνωσης των διαφόρων υπηρεσιών μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας και υπό το φως των νέων διαπραγματεύσεων. Εχθές σας το είχα πει ότι θα προσθέταμε ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων έλαβε την εντολή να συντάξει μία έκθεση για τα εξωτερικά γραφεία της Ένωσης, όπως ε, θα διαμορφωθούν μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Αποφάσισαν λοιπόν ε, στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να κάνουν μία έκθεση για όλα αυτά. Η ΑΦΚΟ λοιπόν θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα του Ιρλανδικού, έπρεπε να περιμένει το αποτέλεσμα του Ιρλανδικού δημοψηφίσματος πριν ξεκινήσει τη διαδικασία για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Είναι ιδιαίτερα ε, στενό το χρονοδιάγραμμα. Η συζήτηση θα γίνει αύριο στην ΑΦΚΟ και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 8 Οκτωβρίου και η έκθεση θα εγκριθεί στις 19 Οκτωβρίου στην Επιτροπή για να υποβληθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε τη γνώμη μας σε ένα θέμα το οποίο επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής δομής της Ένωσης, αποφάσισαν οι συντονιστές να με ορίσουν εισηγητή γνωμοδότησης ως πρόεδρο της Επιτροπής και τους ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η όλη συζήτηση και το πόσο σημαντική είναι η δημιουργία μιας τέτοιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εξωτερική δράση. Η πρόταση έχει σαν στόχο τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εξωτερική δράση, ούτως ώστε να υποστηρίξει τον ύπατο αρμοστή της Ένωσης για τα εξωτερικά θέματα και την πολιτική ασφάλειας, που θα συνδυάζει τους ε, ρόλους ε, ε, του τωρινού ε, είπα του ε, αρμοστή του κυρίου Σολάνα και της Επιτρόπου Εξωτερικών Σχέσεων της κυρίας Φερέρο Βάλνερ. Βέβαια αυτό το θέμα των αρμοδιοτήτων ήταν και το λιγότερο επίπονο ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Όμως η συνθήκη της Λισαβόνας είναι σχετικά ασαφής για το πώς θα ε, στηθεί αυτό το νέο σύστημα. Και έχει μείνει απ' έξω το κοινοβούλιο, το έχουν παραμερίσει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας με την πρωτοβουλία των συναδέλφων της ΑΦΚΟ, ούτως ώστε να συμμετέχουν στη συζήτηση και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης. Για την Επιτροπή Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντική η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας είναι ζωτική σημασίας ούτως ώστε η συνεργασία και η ανάπτυξη να συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν πολιτικώς αυτόνομα με δικούς τους στόχους. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικότατο να έχουμε μια σαφή θέση σε αυτή τη συζήτηση και να εισακουστεί και η φωνή μας κατά τη γνώμη, στη γνωμοδότησή μου μάλλον, εγώ συγκέντρωσα την προσοχή μου στα ουσιαστικά ζητήματα της συζήτησης ε, για την ανάπτυξη και δεν εκφράστηκα για άλλα θέματα ουσίας, δηλαδή ποιο είναι το μέγεθος ε, της υπηρεσίας, ε, αν θα είναι μία απλή γραμματεία του είπα του αρμοστή ή αν θα είναι μία υπηρεσία που θα συσπηρώνει όλες τις γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν για εξωτερική πολιτική και τι ισορροπία θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ της διακυβερνητικής και κοινοτικής διάστασης σε αυτή τη διάρθρωση. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά διαβάζοντας ε, το σχέδιο έκθεσης ε, του Έλμαρ Μπρόκ ε, έχω εμπιστοσύνη στους συναδέλφους της ΑΦΚΟ και της ΑΦΕΤ ότι θα προασπίσουν τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν εγώ συγκέντρωσα την προσοχή μου ε, στο πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα της άσκησης της πολιτικής συνεργασίας και ανάπτυξης, έτσι όπως ορίζεται από τη συνθήκη. Θα βρείτε λοιπόν εσείς ε, στο κείμενο όλους τους όρους που θέτω για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ασκούμε την αναπτυξιακή πολιτική. Θα σας δώσω το λόγο για να κάνετε και εσείς τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων και συμμετείχα σήμερα το πρωί στη συζήτηση σε αυτήν την Επιτροπή για αυτό το θέμα. Δηλαδή τη σύσταση της εξωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα χρόνου, όπως είπε και η Πρόεδρος. Πρέπει εμείς να γνωμοδοτήσουμε ως Κοινοβούλιο πριν αρχίσει να λειτουργεί ο όλος μηχανισμός διορισμού του ΙΠΑ του ε, αρμοστή για την εξωτερική πολιτική και πριν αρχίσει να συγκροτείται η υπηρεσία εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει ως Κοινοβούλιο να ζητήσουμε κάτι το ισοδύναμο με τις ακροάσεις ε, των ε, νέων επιτρόπων. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή του είπα του αρμοστή έτσι όπως ορίζεται η φυσιογνωμία του στη Νέα Συνθήκη της Λισαβόνας. Σε αυτήν την επιτροπή έθεσα και ακολουθώντα και τη γραμμή της Προέδρου δηλαδή ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι μια σημαντική πλευρά της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το 60% της πολιτικής, ε, της αναπτυξιακής πολιτικής ανά τον κόσμο το, το ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ό,τι έχει να κάνει με πολιτικό διάλογο, εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμεύονται άμεσα με την ανάπτυξη. Και νομίζω ότι ακολουθούμε την ίδια γραμμή και οι δύο επιτροπές. Δηλαδή η δική μας και οι συνταγματικών υποθέσεων. Είναι να διατηρηθεί η αρμοδιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής αυτόνομα. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική που γίνεται σε επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας και η γενικότερη εξωτερική πολιτική να λειτουργούν εναρμονισμένα μεν, αλλά να μην καπελώνεται η αναπτυξιακή πολιτική από τον ύπατο ε, αρμοστή για τα εξωτερικά ζητήματα. Συνεργασία λοιπόν, αλλά όχι εξαφάνιση της δικής μας πολιτικής. Μόνο και μόνο δηλαδή για να επεκταθούν οι αρμοδιότητες του είπα του αρμοστή. Ευχαριστώ κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εσείς έχετε στην έκθεση, στο σχέδιο έκθεσή σας επιμείνει πολλές φορές στην αυτονομία της ε, συνεργασίας και της αναπτυξιακής πολιτικής. Πολύ σημαντικό λοιπόν όλο αυτό και θα πω κάτι το θεμελιώδες. Σύμφωνοι με το συντονισμό των πολιτικών. Αλλά δεν θα πρέπει η πολιτική ανάπτυξη και συνεργασίας δεν θα πρέπει να είναι υπόλογη στην εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, άμα εμείς θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια χρηστική δράση και τη θέσουμε υπό την εξωτερική πολιτική, πλέον δεν υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι ένα ανθρώπινο δικαιώματα. Και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε κριτηρία τακτικού ή στρατηγικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να προσθέσουμε λοιπόν μερικά στην έκθεσή σας που να λέει ναι, ότι θα πρέπει να μην ισχύσει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πριν από μερικά χρόνια κατάργησε το Συμβούλιο για αναπτυξιακά ζητήματα. Τότε πρόεδρος του Κοινοβουλίου ήταν ο κύριος Κόξ και εγώ του είχα τηλεφωνήσει και είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Όπως επίσης και αντιρρήσεις είχαν εκφράσει και ορισμένοι πρωθυπουργοί τότε. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία θεσμική αυτονομία στο Συμβούλιο των Υπουργών Ανάπτυξης. Εντάσσεται βέβαια αυτό το ζήτημα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, στο Συμβούλιο Εξωτερικών, και το Συμβούλιο Ανάπτυξης εντάσσεται μέσα στις γενικές υποθέσεις. Έχουν βέβαια τη δική της σχετική αυτονομία, αλλά προς τα έξω φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το Συμβούλιο. Και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και για να το πω δηλαδή ομά, ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίστηκε το θέμα ήταν πραγματικά πολύ χαμηλό προφίλ. Ε, πρέπει εμείς να επανέλθουμε στο ζήτημα και να το βροντοφωνάξουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ευτυχώς που η Σουηδία προεδρεύει, που είναι μια πρωτοπορία σε θέματα απασχόλησης, οπότε ελπίζω ότι η Προεδρία θα μας εισακούσει στις επιθυμίες μας. Euh, Εάν σε άλλους επιθυμεί να λάβει το λόγο, να σας υπενθυμίσω πως μπορείτε να καλυθέσετε τροπολογίες έως την 9 Οκτωβρίου το μεσημέρι, 12.00. Nous attendons, monsieur... Euh, Αναμένουμε τον κύριο Βίλνταρ Χέγκερσεν από το ΙΔΕΑ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή, αλλά προηγουμένως να εξετάσουμε τα δύο τελευταία σημεία της μεσαίας διατάξεως. Σημείο 19. Υπό τα διάφορα υπάρχει κάτι. Αν έχετε κάτι, αυτή είναι η στιγμή. Όχι, πάμε παρακάτω. Η προσεχή συνεδρίασή μας ε, θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου από τις 3 έως τις 30 το απόγευμα εδώ στις Βρυξέλλες και την 3 10 Νοεμβρίου 9 έως 10 και 10 έως 30 αλλά και 3 έως 30 το απόγευμα πάντα στις Βρυξέλλες. Διακόπτουμε λοιπόν ε, μέχρι να αφηχθεί ο κύριος Βιντελ Χέγκερσεν, άρα μέχρι τις 4, 20 λεπτά διάλειμμα. Προλαβαίνουμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Nous euh, la session. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας, να εξετάσουμε τώρα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση του, της δημοκρατίας. Την παρουσίαση μα μας την κάνει η IDEA International πάνω στο θέμα της οικοδόμησης δημοκρατίας και της ε, εκλογικής ε, συνδρομής. Ε, αυτό το Ινστιτούτο εδρεύει στη Σουηδία και κάνει μία μελέτη σε βάθος, σε πάρα πολλούς κλάδους, ε, προκειμένου να προσδιορίσει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα οικοδόμησης της δημοκρατίας. Παρουσίασαν τα ευρήματά τους τον Ιούλιο στην Σουηδική Προεδρία. Το θέμα αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Σουηδική Προεδρία. Η Επιτροπή μας, συγχρόνως με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε προετοιμάσει μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές μας σχέσεις και αυτό για την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Σήμερα έχουμε μεταξύ μας τον κύριο Βίνταρ Χάγκελσεν που είναι γενικού γραμματέας της International Idea και θα μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ε, ομάδας του, του οργανισμού του και θα μας εξηγήσει πώς ε, θεωρείται, ε, πώς εκλαμβάνεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το θέμα της οικοδόμησης δημοκρατίας. Πρώτον να δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Χέγγελσεν. Θα ήθελα η κυρία Χαουτάλα, πρόεδρος της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων να μας πει δύο λόγια. Αλλά δεν έχει ακόμα αφιχθεί. Αυτό σημαίνει πως θα της δώσουμε το λόγο, θα δώσουμε το λόγο αφού θα έχουμε ακούσει την παρουσίαση του κυρίου Εγγελσόνα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Έγγελσεν. Παρακαλώ, ελπίζω να μας εμπνεύσετε με τις, με τις ιδέες σας. Έχετε το λόγο. Thank you uh, very much, Madam Chair, and thank you. Παρακαλώ, ακούγεται η ελληνική δερμηνία. Αν ακούτε ελληνική δερμηνία, την είναι να κάνει ανέβουμε στην καμπίνα υπαριθμών 7. Είμαστε στη διάθεσή σας. Καμπίνα υπαριθμών 7, παρακαλώ. Νομίζω ότι έχει... Nationality as Norwegian, I'm very happy to see a Norwegian represented in the European Parliament. The uh, report that έκθεση που θα παρουσιάσουμε, την έχουμε ήδη παρουσιάσει, σήμερα την παρουσιάζουμε και εδώ, είναι η έκθεση που στηρίζεται στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικοδόμηση της δημοκρατίας. Την έκθεση θα τη διαθέσουμε στα μέλη. Αρχίζω την παρουσίαση με κάποιες βασικές πληροφορίες. Το σκεπτικό, αν θέλετε, που οδήγησε στο εγχείρημα αυτό αρχίζοντας με την κατάσταση της δημοκρατίας παγκοσμίω και την ε, υποστήριξη της δημοκρατίας. Μετά θα αναφερθώ στα συμπεράσματα της έκθεσης, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις και μετά θα κάνουμε ε, συζήτηση. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχους έχουν περάσει χρόνια μετά τις εκλογές, μετά το τέλος του Η τον εκδημοκρατισμό της Λατινικής Αμερικής. Εν πολλής ε, είναι ένα έτος αυτό που οδηγεί σε ε, στοχασμό. Ε, η εικόνα είναι μεικτή. Τώρα τα της δημοκρατίας είναι καλύτερα από ό,τι πριν από 20 χρόνια σε σχέση με πέντε χρόνια και σήμερα, εκεί δεν είμαστε τόσο βέβαιοι για την πρόοδο. Πάντως, ε, ε, η δημοκρατία ζητείται από τους λαούς, το δείχνουν οι στατιστικές, τα βαρόμετρα και βλέπουμε βέβαια και τις αντιδράσεις του κόσμου στη Βερμανία, την Τεχεράνη για παράδειγμα, το καλοκαίρι, υπάρχουν ε, χώρες όπου σημειώνεται πρόοδος στην εκδημοκρατισμό, στην Ινδονησία, πέρσι, στην Κάνα, έγιναν εκλογές ε, ειρηνικές, έγινε μετάβαση της εξουσίας με τρόπο ειρηνικό. Υπάρχουν λοιπόν ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν πρόοδοι. Όμως υπάρχουν και συνεχιζόμενα καθεστώτα αυταρχικά. Πολλά στον αραβικό κόσμο και υπάρχουν και υποτροπές. Ε, στο Ζιμπάμπουε, η Κένια ε, και ώρες τα τελευταία χρόνια και στρατιωτικά πραξικοπήματα που θεωρούσε, θα θεωρούσε κανείς ότι ε, είναι στοιχείο του παρελθόντος υπάρχει στην Ονδούρα στη... και σε άλλες χώρες. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου συγκρούσεις εύθραυστες καταστάσεις καταδεικνύουν τη δυσκολία του να υπάρχουν δημοκρατικές ρίζες στο Αφγανιστάν, στο Σουδάν κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια εικόνα μεικτή. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις που τονίστηκαν ε, στη διεθνή κοινότητα υπάρχουν και σιωπηρές περιπτώσεις δημοκρατιών εύθραυστον, όπου υπάρχει μάλλον μία τυπική δημοκρατία, αλλά η πολιτική διαδικασία δεν είναι τόσο δημοκρατική. Μπορεί να υπάρχει, ας κυριαρχία μονοκομματική, όπου υποτίθεται ότι υπάρχουν ελεύθερες εκλογές, αλλά υπάρχει διαφορά στην πολιτική. Ε, πολλές φορές είναι διεφθαρμένα δύναμα τα πολιτικά κόμματα, δύναμη η αντιπολίτευση έντονη πόλωση στην πολιτική κουλτούρα, συχνές συνταγματικέ αλλαγές, τροποποιήσεις και συχνή χρήση δημοψήφισμάτων που μπορεί να χρησιμοποιούνται σε εργαλεία σε τέτοιες πολλωμένες καταστάσεις. Όλες τις ε, περιπτώσεις αυτές τις χαρακτηρίζει η ε, ικανότητα ή η ανικανότητα της δημοκρατίας να ανταποκρίνεται σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και αυτή η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ανάπτυξης και πώς η υποβοήθηση της δημοκρατίας και της ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει σε αυτά τα πλαίσια είναι στην καρδιά των διεθνών προβληματισμών και διαβουλεύσεών μας. Η ανάπτυξη της δημοκρατίας είναι ρευστή σήμερα. Βλέπουμε ότι αμφισβητούνται παραδοσιακές προσεγγίσεις ε, της, μέσα από τη βοήθεια στην Κίνα, οι ασιατικές τίγρεις αμφισβητούν την δημοκρατία ως βάση ανάπτυξης. Και τα, τις τελευταίες ε, δεκαετίες ε, βλέπουμε ότι ε, σε κράτη όπως το Ιράκ η, δημιουργείται πόλωση και τώρα ενδεχομένως θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Ε, ένα παράδειγμα τέτοιας προσπάθειας είναι η ομιλία του Προέδρου Ομπάμα στο Κάιρο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη μεγαλύτερη οικονομία, είναι ο μεγαλύτερος ε, πάροχος βοήθειας και να κέντρο με ειδικό βάρος ε, διεθνώς μπορεί λοιπόν να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ίσως ε, να είναι... Ε, να μην είναι πολύ δυναμική σε το μίσο ε, στρατιωτικού ενδεχομένω, αλλά έχει μεγάλη ελκτική δύναμη. Και γι' αυτό διεθνώς ε, θεωρήθηκε ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Σουηδία που έχει και την Προεδρία τώρα έθεσε στην αναπτυξιακή συνεργασία ε, στο επίκεντρο την ε, δημοκρατία. Και εμείς ε, προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε να αναλυφθεί μια πολιτική πρωτοβουλία από τη Σουηδία και να κάνουμε διαβουλεύσεις σε όλο τον κόσμο για να δούμε πώς οι άλλες περιφέρειες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη δημοκρατία και την ανάπτυξη. Το, αυτό, το προσφερ, προσφερθήκαμε να το κάνουμε. Είμαστε μια οργάνωση 25 κρατών μελών δημοκρατικών από όλα, όλες τις και έχουμε και δίκτυα και εταίρους σε άλλες περιφέρειες για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους πόρους που υπάρχουν τις απόψεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κάναμε αυτό γιατί αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την πόλωση και το να διέξω το πολιτικό διάλογο για τη δημοκρατία στα διεθνή βήματα, θα πρέπει να μην γίνεται εν κενό η λήψη των αποφάσεων και θα πρέπει να υπάρξει ένας ζωντανός διάλογος πριν από τις πολιτικές αποφάσεις, ώστε να υπάρχει διάλογος, να υπάρχουν επικοδομητικοί όροι. Ε, γι' αυτό αρχίσαμε διαβουλεύσεις διεθνώς ε, σε όλο τον κόσμο ε, και όλα αυτά οδήγησαν, κατέληξαν στην έκθεση αυτή η οποία καταλήγει σε τέσσερα συμπεράσματα τα οποία θα σας παρουσιάσω. Καταρχήν, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιτυχής. Αν ακούσετε συζητήσεις στην Ευρώπη, στους κόλπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκεί στους περίκους, στους παρικούντες, θα δείτε πολλές φορές ένα ζωφερό κλίμα, επικεντρώνονται στις δυσκολίες. Ενώ έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κόσμος βλέπει ως πολύ επιτυχημένη την Ένωση και υπάρχει μια επιθυμία να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφηγείται την ιστορία αυτή. Πώς τα κατάφεραν τόσο καλά. Δηλαδή, πώς μπόρεσε πάνω στις στάχτες των πολέμων και των καταστροφών να χτίσει ε, μια ε, περιφέρεια ε, που ευημερεί με οικονομικό δυναμισμό, με κοινωνική συνοχή κλπ. Τι πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα μέσα στις χώρες και μεταξύ χωρών και ήταν κύριοι, κύριες κινητήριες δυνάμεις για την πρόοδο αυτή. Είναι μια εμπειρία ενότητας, μια εμπειρία διαφορετικότητας που πρέπει να ε, μεταλαμπαδευτεί κι αλλού. Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόσει το εξωτερικό αυτό που εφαρμόζει το εσωτερικό. Όταν ο κόσμος ε, κοιτάζει την Ευρώπη, βλέπει μία ήπειρο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι σεβαστά, όπου δεν επικεντρώνονται μόνο στα, οικονομικά, στα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Βλέπουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ε, όχι μόνο τύπης, αλλά και σε μια ουσιαστική δημοκρατία η οποία αποδίδει. Είναι μια ευρύτερη, συνολικότερη άποψη για τη δημοκρατία αυτή. Άλλες χώρες, άλλες περιοχές βλέπουν τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, τις βιώνουν. Μέσα από εκεί βλέπουν μια πιο στενή εφαρμογή της δημοκρατίας και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της δημοκρατίας βλέπουν έμφαση στις εκλογές, για παράδειγμα, κυρίως ε, παρατήρηση των εκλογών. Δεν βλέπουν πώς στις εξωτερικές δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τις επιτυχημένες συνταγές, αν θέλετε, που δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει μια μεγάλη επιθυμία να το δουν αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση, συνεκτική και εταιρική σχέση για την οικοδόμηση της δημοκρατίας παντού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι μια επιθυμία να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ισχυρότερη σε θέματα δημοκρατίας, ακόμα και σε περιοχές όπου δεν θα περίμενε κανείς ότι θα ήθελαν πιο ισχυρά μηνύματα, υπάρχει επιθυμία να εμένει στις αρχές της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλές γωνιές του κόσμου θεωρείται ως ε, εμπόδιο για το, το εμπόριο. Ε, πολλές φορές ε, την διαφοροποιούν από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουν στις αρχές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από, ε, σε όλα τα επίπεδα ε, και να μην ε, περιορίζεται στο ρόλο της ως ας πούμε ένα εμπορικό κέντρο μια ομάδα χωρών που ασχολείται με το εμπόριο. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό οι εταίροι μέσα από ενημέρωση, διαβούλευση, άνοιγμα, διαφάνεια. Υπάρχει επίσης προβληματισμός για τα διπλά μέτρα και σταθμά. Και στον αραβικό κόσμο ακούσαμε το θέμα των εκλογών στην Παλαιστίνη να ε, συζητείται ξανά και ξανά. Και βέβαια είναι σημαντικό ότι υπήρχε, θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση ενιαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχε των μεμονωμένων χωρών. Είναι σημαντική πρόκληση αυτή η οποία ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της, ε, ε, των εκκλήσεων από την Ευρώπη για ελεύθερες εκλογές και δημοκρατία. Το τέταρτο και τελευταίο κύριο συμπέρασμα είναι μια έκκληση για γνήσιες εταιρικέ σχέσεις, για γνήσιο διάλογο. Ίσως και για κάποια μετριοπάθεια ταπεινότητα, σεβασμό του γεγονότος ότι πολλοί έρχονται με διαφορετικό υπόβαθρο, ιστορία, ε, πλαίσιο, κουλτούρα αν θέλετε. Ε, υπάρχουν διαφορετικά ε, δεδομένα στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να γίνει σεβαστή η διαφορετικότητα σε όλες τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλο τον κόσμο πρέπει να εγκαταλείψουμε τη σχέση δωρητή παραλήπτη και να υπάρχει μια γνήσια εταιρική σχέση. Και η γλώσσα της προώθησης της δημοκρατίας θα πρέπει να αντικατασταθεί μέσα από συνεργατική οικοδόμηση της δημοκρατίας, ούτω ώστε να υπάρχει πιο ισότιμη ε, σχέση, σχέση ίσου προς ίσον στην προαγωγή της δημοκρατίας και την υποστήριξή της. Και αυτό το τελευταίο συμπέρασμα ε, έχει σχέση με τις παρατηρήσεις που θα ακολουθήσουν τώρα σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Ποια θα είναι τα σημαντικά επόμενα βήματα. Καταρχήν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον διάλογο. Αυτό που βλέπουμε όταν ανοίγουμε συζητήσεις σε όλο τον κόσμο, όπου καλούνται οι χώρες και οι περιφέρειες να δουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν περιορίζονται εκεί, αλλά κάνουν και ε, κριτικές παρατηρήσεις και συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση στη δική τους περιοχή. Αυτό το κάνουν γιατί αναγνωρίζουν ε, ότι εδώ υπάρχει ένα γνήσιο ενδιαφέρον ισότιμο ενδιαφέρον για τον διάλογο. Και όχι μόνο υπάρχει ενδιαφέρον για συνέχιση και προαγωγή του διαλόγου, αλλά υπάρχει και μια επίσημη βάση με τον, τη χάρτη για τη δημοκρατία, σε διάφορες περιοχές και ο νέος χάρτης ΑΣΕΑΝ έχει αναφορές κάπως αδύναμες στη δημοκρατία και ε, σε άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν τέτοιοι χάρτες παρόλα αυτά γίνονται ζωντανές συζητήσεις για θέματα δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν ένα συμπέρασμά μας είναι ότι στον τομέα της δημοκρατίας και της ανάπτυξης θα πρέπει να υπάρξει συνεχιζόμενος διάλογος μεταξύ περιφερειακών οργανώσεων για τις προκλήσεις, για τις δυνατότητες που ανοίγονται από τα μέσα αυτά και πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μέσα από σχέσεις εταιρικέ. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη υποστήριξη από την Ένωση της Δημοκρατίας, καλύτερες συνέργειες μεταξύ δημοκρατίας, ανάπτυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ε, ε, δημοκρατίας και της Ανάπτυξης, η Προεδρία του του Συμβουλίου πήρε την πρωτοβουλία για να διαμορφώσει καλύτερα τις πολιτικές αυτές και τα, ο σκοπός είναι να καταλήξουν σε συμπεράσματα του Συμβουλίου. Χαίρομαι που βλέπω την ε, προφορική ερώτηση της Επιτροπής σας και χαίρομαι διότι και άλλες επιτροπές και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, συνεργάζονται γιατί αυτό χρειάζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιηθούν οι προφορικές ερωτήσεις και η συνέχεια που θα δοθεί σε αυτές στο έπακρο. Επίσης, ε, δύο κύρια συμπεράσματα είναι να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή εμπειρία και δεύτερον να εφαρμοστεί μια ευρεία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημοκρατία που μπορεί να δει με κριτικό μάτι επιμέρους περιπτώσεις αλλά έχει και μια προοπτική ε, μακρότερης Και τέλος θα πρέπει να γίνει πιο ζωντανή η δημοκρατία, να ζωντανέψει και μέσα από τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε αυτό το τομέα θα παίξουν μεγάλο ρόλο οι βουλευτές οι οποίοι έχουν να λογοδοτούν προς τους εκλογείς και γι' αυτό πρέπει να είναι οι πρεσβευτές που θα συνηγορήσουν υπέρ μιας καλύτερης μακροπρόθεσμης ε, προσέγγισης σε θέματα οικοδόμησης δημοκρατίας. I now give the floor to Mrs. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Πρόεδρος της ε, Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, που μας ζητήσατε να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι εκεί η εξέταση του ζητήματος και ευγνώμων για την ευκαιρία που μας προσφέρετε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την έκθεση που συνέταξε η ΑΙΔΙΑ σχετικά με τις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εκδημοκρατισμού διότι για μας έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε πως οι καλές μας προθέσεις δεν γίνονται αντιληπτές παντού με τον ίδιο θετικό τρόπο. Ειδικά θα πρέπει να αποτανθούμε σε αυτούς που θέλουμε εντό εισαγωγικών να εκπολιτήσουμε. Καλό είναι να ακούγεται πως θα πρέπει να διηγηθούμε την επιτυχή ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακαλώ διορθώστε με αν υπερβάλλω, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη διεθνική οργάνωση που θέλει να καταστεί απόλυτα δημοκρατική. Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι ακόμα δεν είμαστε μια τέλεια δημοκρατία, αλλά θα το πετύχουμε. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε με διάφορους θεσμούς και το οργανισμό σα, το IDEA, θα είναι ένας πολύ καλός εταίρος. Στην υποτρίωτη του δικημάτου έχουμε το προνόμιο να δουλεύουμε με το Ινστιτούτο της Βενετίας και το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο για τον εκδημοκρατισμό που είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν 41 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και εμείς ε, χρειάζεται να συζητάμε περισσότερο με τους ερευνητές αλλά και οι ερευνητές επιθυμούν να συζητούν μαζί μας διότι τα πράγματα είναι όπως και ο κόσμος ιδιαίτερα περίπλοκα. Λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις σα αναφορικά με το θέμα της τη δημοκρατίας και εγώ το προνόμιο να, συν, που συνάντησα την κυρία Κρίστενσεν σήμερα το πρωί και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ καλά προσδιορισμένα και μπορούμε να αναφερόμαστε σε κάποια νομικά κείμενα. Αλλά το αυτό δεν συμβαίνει με τη δημοκρατία. Μπορούμε να έχουμε συζητήσεις ε, πολύ ωραίες ε, σχετικά με το δημοκρατία και πρέπει να διεξαχθούν αυτές οι συζητήσεις. Ε, έχουμε τους ορισμούς μας, αλλά φυσικά δεν θα πρέπει να δούμε τον εκδημοκρατισμό ως μια απλή βοήθεια προς τις χώρες ε, να οργανώσουν εκλογές. <clears throat> και μια ερώτηση που θα ήθελα να θέσω θα πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο της δημόσιας συμμετοχής περισσότερο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αναφέρουμε σε ένα ε, νομικό μέσο που ονομάζεται η Σύμβαση του Άρους που δίνει στους πολίτες πολλών κρατών την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αφορά το θέμα αφορά γενικά το περιβάλλον, αλλά εδώ μπορούμε να προωθήσουμε τα συμμετοχικά δικαιώματα των πολιτών. Και η ερώτησή μου είναι εξή. Έχετε εργαστεί επί της ε, επιθεμάτων συμμετοχής, διότι αυτό αποτελεί και το κλειδί για να δώσουμε φωνή στους ε, πληθυσμούς ε, των φτωχών και φτωχότερων χωρών προκειμένου να μπορούν να εκφράσουν αυτά τα οποία προσδοκούν από τους ε, πολιτικούς και από τους καταρτίζοντες ε, την πολιτική δράση. Με ιδιαίτερη χαρά άκουσα από τον κύριο Βέτερ ε, ότι η ιδέα είναι από τον κύριο Βίταρ, Η πρόθεσή μας είναι να αποθήσουμε την δημοκρατία και η Εύα Τζολή και άλλοι επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στις παρόμοιες συζητήσεις εάν και εφόσον μας προσκαλέσετε. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκερέρα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την παρουσίαση αυτής της μελέτης του IDEA International ε, εμπειρογνώμων τόνισε πως αν ε, συγκρίνουμε την ισχύουσα κατάσταση με αυτή που υπήρχε πριν από τρία κονταετία, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα πως η δημοκρατία έχει προοδεύσει σημαντικά κατά τη διάρκεια αυτή τη τρία κονταετία. Αν όμω κάνουμε σύγκριση με τα τελευταία πενταετία, τότε έχουμε κάποιε εμβολίες αναφορικά με την σταθερότητα των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Το βέβαιο είναι πως ε, αυτές τις στιγμές του 21ου αιώνα το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε δημοκρατίες ε, είναι γύρω στο 40%. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες όπως το Human Rights Watch και αυτό το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στις, ε, στον 20ο αιώνα. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι της, της ανθρωπότητας 100 χρόνια αργότερα συνεχίζει να ζει υπό μη δημοκρατικά καθεστώτα. Ένας ε, ε συγγραφέας ο Τζον Ντάν ε, ε, έχει γράψει ένα βιβλίο του ότι η δημοκρατία αποτελεί ένα ημιτελές ταξίδι. Δεν είναι ένα ημιτελές ταξίδι, αλλά είναι ένα ταξίδι με διακοπές και συχνά με οπισθοδρομήσεις. Θεωρώ πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επιτυχής Ήπειρος μια επιτυχημένη ιστορία και έχουμε διδάγματα τα οποία πρέπει να διδάξουμε και να καταδείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Παραδείγματο χάρη είναι μια κοινωνία όπου είναι συχνός ο διάλογος ο πλουραλιστικός, όπου υπάρχουν κοινωνικές συμφωνίες, όπου έχουμε πολιτικές συνοχής και υπάρχουν διαδικασίες συνενετικές. Θεωρώ λοιπόν πως ε, θα πρέπει να όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά με ανησυχεί κάτι που ανέφερε ο εμπειρογνώμονά μα, ότι δηλαδή χρειάζεται να το... Δεν πρέπει να το πράττουμε με αλαζονία ή με αυταρέσκεια. Ο Μπίρχου Πάρεκ, ένα άλλο μελετητή τη δημοκρατία, ε, καθόρισε πως υπάρχουν κοινωνίες ε, στον κόσμο που δεν ε, λειτουργούν με έννοια του κτητικού ατομικισμού που είναι τα χαρακτηριστικά της, των πλουρανιστικών δημοκρατιών της Δύσης. Οι εμπειρογνώμονας μας σε ανθρώπινα δικαιώματα μόλις μας είπε διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε δίκαιο και δημοκρατία τα δικαιώματα είναι σωστά προσδιορισμένα, οι δημοκρατίες όμως ε, οικοδομούνται από πολιτιστική σκοπιά. Υπάρχουν λοιπόν πολλές περιοχές στον κόσμο όπου αυτοί δρούν περισσότερο τα θεσμικά όργανα και ο κολεκτρισμός Χρειάζεται λοιπόν να μην ε, δείξουμε αναλγησία στα χαρακτηριστικά των υπολείπων κοινωνιών. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στις ε, αξίες μας, ειδικά όταν θελήσουμε να τις ε, καταδείξουμε και να τις μεταλαμβαδίσουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Τόσο από πλευράς εκτελεστικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Thank you. Ευχαριστώ. Η Σουηδική Προεδρία θέλει να πει κάτι. Η Κομισιόν μήπως. Ούτε. Δεν μας μένει παρά να ευχαριστήσουμε τον ιδέα για τη συμμετοχή του και τη συνεισφορά του. Θα σημειώσουμε, να βάλουμε υπόψη μας μάλλον όλες τις συστάσεις τους. Εξετάσαμε και πριν από λίγο τα δύο τελευταία σημεία. Τελειώνει λοιπόν η συνεδρίασή μας για σήμερα. Λοιπόν, θα σας δώσω την αίθουσα. Είναι η αίθουσα 2Q2. Θα συναντηθούμε λοιπόν, εκεί με την ΑΦΕΤ για τη διανομή των γραφείων Ζαχάροφ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.